κοινωνική ευθύνη ακόμη και στις εμπορικές ε, συμφωνίες πρέπει να είναι δυναμική και να προσαρμόζεται όταν πρέπει να καλύψουμε και άλλους τομείς. Ευχαριστούμε κυρία Μπερές. Δυο μισή λεπτά από την Κοινωνική Επιτροπή. Σαν εισηγητής